Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η δήλωση της Επιτροπής για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Σήμανσης. Είναι ένα σημείο το οποίο βέβαια είναι πολύ επίκαιρο δυστυχώς, γιατί ακριβώς εδώ στις Βρυξέλλες πριν από λίγες μέρες έλαβε χώρα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα για το οποίο βέβαια θα συζητήσουμε μια που έχουμε αυτό το θέμα. Θέλω να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα, στις οικογένειές τους. Καλωσορίζουμε εδώ για τη συζήτηση τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Σιμ Κάλλας, τον Επίτροπο. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα στην Κορούνια συζητούσαμε μαζί για θέματα ασφάλειας στη θάλασσα. Και μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και σε βάθος συζήτηση εδώ για την Αλία. Οπότε συνεχίζουμε τώρα λίγο πολύ στο ίδιο νήμα που συνδέει τα δύο θέματα. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον Επίτροπο, τον ε, κύριο Κάλλας, για να μας κάνει τη δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά το θέμα αυτό της ασφάλειας των σιδηροδρόμων που θα μας απασχολήσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε να ανοίξει έτσι η συζήτηση αυτή. Το ατύχημα στο Μπάζιγκεμ πριν από λίγες μέρες φυσικά και ήταν μια φοβερή τραγωδία. Μετά από αυτό το σοβαρό ατύχημα σίγουρα τίθενται πολλά τεχνικά και πολιτικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, η σκέψη μας βέβαια είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να βρει κανείς λόγια παρηγορητικά μετά από τόσο σοβαρά ατυχήματα. Μερικέ φορέ η σιωπή λέει περισσότερα. Οι αιτίε δεν είναι απόλυτα γνωστέ και οι τεχνικέ έρευνε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται σύμφωνα με τι διατάξει τη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ασφάλεια. Είναι ευθύνη των ε, βελγικών αρχών να φέρουν σε πέρα στην έρευνα αυτή, η οποία πρέπει να λάβει χώρα ανεξάρτητα φυσικά. Ο στόχος δεν είναι μόνο το να βρούμε τον υπεύθυνο, αλλά να βρούμε επίσης και τρόπους για να βελτιώσουμε την κατάσταση και να προλάβουμε στο μέλλον τέτοια ατυχήματα. Ζήτησε η Ερευνητική Επιτροπή αυτή και από το Ευρωπαϊκό Αρμόδιο Σώμα, τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών, να βοηθήσει στις έρευνες αυτές και ξεκίνησαν οι έρευνες λίγες ώρες μετά το ίδιο το ατύχημα. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι όσο τα αίτια δεν είναι απόλυτα γνωστά, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Φυσικά και είμαι έτοιμος να εξηγήσω μερικά πράγματα που έγιναν γνωστά μετά το ατύχημα, όπως θέλετε φαντάζομαι. Όπως πολύ συχνά συμβαίνει όταν έχουμε τέτοια ατυχήματα στους σιδηροδρόμους, πολλές φορές μιλάμε για τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ότι αυτοί φταίνε. Πρώτα απ' όλο λοιπόν θέλω να είμαι ξεκάθαρος όσον αφορά την ανοιχτή αγορά. Το άνοιγμα της αγοράς, η ελευθέρωση της αγοράς ε, δηλαδή, επέτρεψε τον ανταγωνισμό και βοήθησε να ξεχωρίσουμε την υποδομή από τη μια μεριά και την επιχείρηση εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων από την άλλη. Αυτό βοηθάει στην ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στους σιδηροδρόμους παραμένει παρόλο που είναι στο κάθε κράτος μέλος να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες. Τακτικά έχουμε εκθέσεις όσον αφορά την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και υπάρχουν ελεγκτές και στα κράτη-μέλη. Οι διάφοροι δείχτες δείχνουν ότι η ελευθέρωση της αγοράς σιδηροδρόμων στον ανταγωνισμό με τίποτα δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις επί της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε ιδέα που συνδυάζει το άνοιγμα της αγοράς με τη μείωση της ασφάλειας είναι λάθος. Η συνύπαρξη τώρα εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων είναι κάτι που βοηθάει. Έχουμε πάνω από 20 διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίζουμε για την ασφαλή διακίνηση των σιδηροδρόμων. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από δύο στοιχεία. Το ένα δίνει πληροφορίες στον υπολογιστή και από εκεί και πέρα ο υπολογιστής φροντίζει για την τροχοπέδηση. Προκειμένου να λειτουργούν τα συστήματα αυτά, με τα τρένα και τις γραμμές, πρέπει να υπάρχει εξοπλισμό συμβατών συστημάτων. Τα επίπεδα ασφάλειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όπως και οι κανόνες πολλές φορές που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό των γραμμών αλλά και των βαγονιών. Η έλλειψη συμβατότητας μεταξύ εθνικών συστημάτων δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τα... τους διεθνείς σιδηροδρόμους γιατί πρέπει να αλλάζουν τα βαγόνια σε κάθε σύνορο αν δεν έχουν τα συστήματα που πρέπει. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν και μέσα στην ίδια χώρα διαφορετικά συστήματα. Το Θαλής, για παράδειγμα, πρέπει να έχει 7 διαφορετικά εθνικά συστήματα, περνώντας από 4 διαφορετικές χώρες. Αν είχαμε ένα ενιαίο σύστημα θα ήταν καλό. Έχει αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα και σιγά σιγά το εγκαθιστάμε σε διάφορα διεθνή τρένα. Το CRDMS που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα διακίνησης σιδηροδρόμων. Πολλά από τα εθνικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί ήδη από τη δεκαετία του 80. Χρειάζεται όμως χρόνος για να τεθούν σε εφαρμογή. Σε πολλές χώρες μόνο ένα μέρος του εθνικού δικτύου ε, εξυγχρονίζεται. Πολλά είναι εδώ και 20 χρόνια έτσι. Υπάρχουν ε, προδιαγραφές από το 2000 πάντως και πολλά πιλωτικά προγράμματα έχουν λάβει χώρα από το 2005 και πολλά, ε, πολλοί σιδηρόδρομοι με το Διεθνές Σύστημα κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές γραμμές. Υπάρχουν ε, πάντως προγράμματα σε όλες τις χώρες μέλη. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, Άχεν Λιέγη. Εκεί υπάρχει μια τέτοια γραμμή και τα σχετικά τρένα είναι εξοπλισμένα με αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει δυνατότητα για τα τρένα να μπορούν να περνάνε τα σύνορα χωρίς να χρειάζονται αλλαγές και θεωρείται και ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την ασφάλεια. Το σύστημα λειτουργεί πλήρως σήμερα, όμως επειδή χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εγκατασταθεί στα τρένα και στις γραμμές και τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, εξακολουθεί το σύστημα αυτό να συνεπάρχει με διάφορα εθνικά συστήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν πλήρης διαλειτουργικότητα. Το σύστημα είναι σίγουρα το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά. Πολλά ερωτήματα τίθενται όταν συγκρίνουμε την κατάσταση αναχώρα. Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε με μια ιεράρχηση, ένα κατάλογο που να βάλουμε τις χώρες. Εξαρτάται κάθε φορά από το τι δείκτες χρησιμοποιεί κανείς, ποια είναι η περίοδος αναφοράς και ποιες είναι οι ποιοτικές εκθέσεις που έχουμε. Σίγουρα τα ατυχήματα επηρέαζουν πάρα πολύ ε, την κατάσταση, όποια και αν είναι η ιεράρχηση που έχουμε φτιάξει μεταξύ των χωρών δεν μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο. Έχει συστήματα προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με τους ομιλητές που μιλάνε καταρχήν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα, από το ΕΛΚ, ο κύριος Ματιέ Γκρός. Για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω και εγώ για τις δηλώσεις σας και ε, μετά το δυστύχημα στο Μπέζιγεν, ε, χρειαζόμαστε να εκφράσουμε τον σεβασμό μας αλλά και το σεβασμό μας προς την έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να προβούμε σε πρώιμα συμπεράσματα ούτε να επιρρύψουμε ευθύνες παρά το γεγονός ότι θεώρησα σωστό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν, γιατί ξέρουμε ότι το θέμα αυτό έχει παραμείνει στο θέμα της εθνικής αρμοδιότητας και αυτό θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το καταδικάσουμε γιατί πρόκειται για ένα θέμα ασφάλειας, ένα θέμα διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων ε, συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κρίμα που δεν είχε δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στο θέμα αυτό στο παρελθόν όπως συχνά γίνεται στην πολιτική. Ε, ακολουθούν εκ των υστέρων οι νέες προτάσεις ε, εγώ θα ήθελα και νομοθετικά να γίνουν προσπάθειες, αλλά και τεχνολογικά, γιατί δεν είχαμε θεωρήσει την, την τεχνολογία αυτή ως τεχνολογία προτεραιότητας, γιατί υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η τεχνολογία εκείνη και θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στο Βέλγιο από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Υπήρχαν λοιπόν δεν υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές. Το μέλλον όμως είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και θα ήθελα να πω ότι για το μέλλον σίγουρα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι καλή εκπαίδευση στον συνδεδομικρό κλάδο. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ε, σχέδια μεταρρύθμισης σε κάθε χώρα. Δεν αρκεί η καλή θέληση. Νομίζω ότι χρειάζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και εδώ, στο Κοινοβούλιο, έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε συγκεκριμένου στόχου. Και μια τρίτη πρόταση εκ μέρου μου θα ήταν ε, η εξή. Νομίζω ότι και οι επιβάτε ε, έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται κατά πόσο η γραμμή την οποία χρησιμοποιούν είναι ε, σωστά εξοπλισμένη. Νομίζω ότι τουλάχιστον χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση των επιβατών για το μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα για δύο λεπτά και μισό έχει το λόγο ο κύριος Ελ Κατραουή. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ξεκινήσω κι εγώ εκ μέρους των σοσιαλιστών με συλληπιτήρια βέβαια για τα θύματα στις οικογένειες των θυμάτων του ατυχήματος αυτού. Περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα της έρευνας για να μπορούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Όμως η ασφάλεια στους σιδηροδρόμους πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς η πολιτική ασφάλειας πρέπει να αξιολογείται τακτικά και όπως και ο συνάδελφος θέλω και εγώ να πω στον Επίτροπο ότι και εγώ λυπάμαι που πολλοί, ακόμα και υψηλά ιστάμενοι στο Βέλγιο, τα βάλανε με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Σήμερα, 2010, στο βελίο όντως είναι εξοπλισμένα τα τρένα μας με τα αυτόματα συστήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να είμαι ειλικρινή, θέλω να πω ότι η ανάπτυξη αυτή τη ωραία ιδέας ενό ε, συστήματο ενιαίου που να αντικαθιστά τα 20 σήμανση, ε, χρειάζεται χρόνο και έχει να κάνει με την τεχνική πολυπλοκότητα. Έχουμε 27 χώρε, όταν ξεκινήσαμε είχαμε λιγότερε, αλλά πάση περιπτώσει όλες οι χώρε πρέπει να συμφωνήσουν με μια ενιαία προδιαγραφή και αυτό έχει δημοσιονομικέ συνέπειε, όπω καταλαβαίνετε. Όπω πολύ σωστά πάντω είπατε, το, η κάθε χώρα θέλει το δικό της σύστημα, αλλά προσπαθούν σιγά σιγά να εφαρμόσουν και το ευρωπαϊκό. Πάντω πρέπει να κοιτάμε μπροστά πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, πώ μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλείς σιδηρογραμμέ. Και αυτό θα το πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω, με το αυτόματο σύστημα RTMS και μην ξεχνάμε ότι το 2009 είχαμε βάλει 240 εκατομμύρια για τα ευρωπαϊκά δίκτυα 10. Έπειτα, Κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων είναι να ελέγξουν κατά πόσο τίθενται σε εφαρμογή κανόνε ασφάλεια. στην πράξη, αν πράγματι γίνεται αυτό. Διότι με τα 10 λέμε ότι πρέπει οι αρχές ασφάλειας σε κάθε χώρα μέλη να έχουν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει την ασφάλεια. προκειμένου πιο συγκεκριμένα η ασφάλεια να προωθείτε, να συντηρείτε και να εξελίσσετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο Βέλιο εγώ δεν νομίζω ότι πάει καλά αυτό, ότι λειτουργεί καλά. Και θα έπρεπε να υπάρξει ένας έλεγχος, με εποπτεία, να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν τις δυνατότητες πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουν ασφαλείς σιδηροδρομικές γραμμές στην επικράτειά τους. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ελκαντραουή. Δύο λεπτά τώρα εκ μέρου των φιλελεύθερων ο κύριος Στέρκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και εγώ εκ μέρου της ομάδας μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Και εγώ θέλω να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να καταλάβουμε τι έφτιαξε. Στη χώρα μου βέβαια γίνονται ζητήματα όσον αφορά την Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει από αυτούς που είπαν ότι εμείς δεν προσέχουμε την ασφάλεια. Ήμουν εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ασφάλεια. Το θυμάται και ο συνάδελφο Ελ Καντραουή, βέβαια. Και ήμουν περήφανο τότε για τη δουλειά που είχαμε κάνει. Και είχα πει τότε ότι οι απαιτήσει μα όσον αφορά την ασφάλεια σε όλε τι χώρε μέλη πρέπει να είναι πολύ υψηλέ. Το είχα τονίσει αυτό. Και με κόπο πετύχαμε να περάσει αυτό από τα κράτη-μέλη. Έγινε όμω. Όντω, σε μερικές χώρες και στη δικιά μου δυστυχώ οι οργανώσεις επιμένουν στην εθνική οργάνωση, η οποία δεν είναι επαρκή. Και ο επίτροπο πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Ίσως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία και να ενισχύσουμε το πλαίσιο, όπω είπε και ο κύριο Γκρό. Γιατί δεν μπορεί η ασφάλεια να μένει πίσω, καθ' άλλο. Έπειτα, όσον αφορά τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται. Τι θα γίνει με αυτούς. Χαίρομαι πάντως που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τον ε, κανονισμό αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που είπαν ότι φταίει το άνοιγμα της αγοράς, η ελευθέρωση της αγοράς. Έτσι μειώθηκε η ασφάλεια. Ε, όχι λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το λέω και επιμένω. Τα στοιχεία που έχουμε από το 2008 από, την, ε, από τον Οργανισμό Σιδηροδράμου είδαμε ότι η Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία πήγανε καλύτερα από όλες τις άλλες που είναι δύο χώρες που άνοιξαν την αγορά τους. Να δούμε τώρα τι λένε και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τομέα, είτε στην ε, διοίκηση, στη διαχείριση, μηχανοδηγή κλπ. Χρειάζονται κατάρτιση, καλή οργάνωση της δουλειάς τους. Αυτά διασφαλίζουν την ασφάλεια. Τέλο, Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι οι σιδηρόδρομοι πρέπει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφοι. Εκ μέλους των Πρασίνων τώρα το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Ιζαμπέλ Ντουιρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Και για μένα το τραγικό δυστύχημα τη περσμένη εβδομάδα είναι η χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή που γνώρισε από το 2001 το Βέλγιο εποχή που ασχολήθηκα προσωπικά όσον αφορά το Υπουργείο Μεταφορών και Κινητικότητας. Ξεφτόμαστε την Κλόβια Διάγκο και τους άλλους, ε, και άλλα θύματα και τους συγγενείς τους και τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο. Και εγώ δεν θα συναγάγω συμπεράσματα τώρα, διότι διεξάγεται η έρευνα και δεν προδικάσουμε τα απορίσματα. Είναι σαφές όμως ότι στο Βέλγιο μπορούμε να κράσουμε τη λύπη μας ότι οι σιδηρόδρομοι άργησαν τόσο πολύ για να καταστήσουν ένα σύστημα αυτόματης προστασίας των σιδηροδρόμων. Και άκουσα την επόμενη της καταστροφής ότι δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για οικονομίες. Και γιατί άργησαν να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Ότι λόγω ελλείψεως χρημάτων δεν εφαρμόστηκαν αυτά και αυτό είναι πολύ πενιχρή δικαιολογία. Και νομίζω ότι έτσι είναι εις βάρος. Το RTMS ε, δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες να επενδύσουν συντονισμένα και δηλειτουργικά στην ασφάλεια θα πρέπει να απαλλαγούμε από τα πολλά εθνικά πρότυπα που θέτουν τροχοπέδι στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα ενώ το STS αναπτύχθηκε, αναπτύχθηκε και θα εξελιχθεί περαιτέρω και πρέπει να υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο τεχνολογικό γι' αυτό. Σε 5-10 χρόνια ακόμα θα έχουμε πολύ περισσότερε εξελίξει. Τέτοια αποτελέσματα, όσο και σπάνια να είναι, πρέπει να, να θυμίσουμε ότι πάντα μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα όσον αφορά την ασφάλεια και θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιε προτάσει. Καταρχά, όπω ξέρετε, κύριε Επίτροπε, συζητούμε για την ώρα τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Ποια θα είναι οι συνθήκε και τα κριτήρια και αυτά. Πιστεύω ότι το RTMS, η χρήση σε όλη την Ευρώπη αυτού του συστήματο ασφαλεία μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Νομίζω ότι και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να θέσουμε και κάποιες προθεσμίες και μέσα υποχρεωτικά μέχρι τότε θα, είναι, θα πρέπει να εφαρμόζονται και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα συστήματα ασφαλεία ταυτόματα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια όσον αφορά τον τομέα τη αγορά. Οι νέοι εμπορευόμενοι που εκμεταλλεύονται στα εθνικά δίκτυα τα τρένα να πρέπει να προσαρμοστούν δεόντω στι προδιαγραφέ ασφαλεία για το σύστημα ταυτόματο ασφαλεία που υπάρχει στα δίκτυα και να εξοπλίσουν ανάλογα και τι ε, ατομηχανέ του και το πλήρωμα να ενημερωθεί και οι σειρμοί να εξοπλιστούν. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να συνδράμει στι προσπάθειε αυτέ για καλύτερη, ε, καλύτερο συντονισμό των εθνικών αρχών ασφαλεία, ούτω ώστε να μπορεί να ε, δίνεται και η αναγκαία άδεια και στον εξοπλισμό των τροχαίων. Ένα λεπτό τώρα. Εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριο Έπινγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματο στον Μπάζουγεμ δεν είναι γνωστά ακόμα. Όμως η διαπίστωση υπάρχει ότι όταν γίνεται ένα τύχημα στην Αγγλία για παράδειγμα λέμε αμέσω ότι φταίει η ελευθέρωση του τομέα. Όμως οι Βέλγοι και οι σιδηρόδρομοι παίρνουν τις περισσότερες επιθετήσεις ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανά επιβάτη και ένα χιλιόμετρο λιγότερα η Γαλλία, 24 cents, ε, η Αγγλία 4 cents κλπ. Παρά τις επιδοτήσεις όμως οι βελγικοί σιδηρόδρομοι έχουν ένα χρέος 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μα τι γίνεται με τα χρήματα, πού πάνε. Αν δούμε τις υποδομές των βέλγικων σιδηροδρόμων βλέπουμε ότι όλα είναι παλιά, απαρχιωμένα. Και τα συστήματα επίσης. Πληρώνεται στους μισθούς, τα χρήματα αυτά πάνε στους μισθούς, πού πάνε. Είναι ένα σοσιαλιστικό τομέα, είναι αλήθεια, στο Βέλγιο, οι σιδηρόδρομοι, με κακή διαχείριση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν λεφτά οι Βέλγοι σιδηρόδρομοι και γι' αυτό είχαν το ατύχημα ή δεν είναι σύγχρονοι. Τώρα ο κύριο Ζακή ένα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τον περασμένο Νοέμβριο σε αυτό το στο ο κύριος Σίμψον δήλωνε ότι το σύστημα του συνδρομικό το κοινοτικό είναι πάρα πολύ ασφαλές και ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι τα τελευταία χρόνια χάρη στην ε, απελευθέρωση της αγοράς. Ε, ε εγώ κόντεψα να πνιγώ με αυτά που άκουσα όμως έγιναν πολλά θανάσιμα ατυχήματα και τίθενται ερωτήματα σε αυτή την ασφάλεια από μετά το ατύχημα του Μπίσιγκεν ήταν ο τελευταίο ο φοβερός απολογισμός από τα θύματα, ψυχολογικά τραύματα που είχαν ε, οι τραυματίες και όλα αυτά μα υπεθυμίζουν ότι είναι και η ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει ε, είναι απρόβλεπτο κάθε αντιστοίχημα βέβαια, αλλά πρώτος παράγοντας ανασφάλειας σε όλα τα συνδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη είναι άμεση συνέπεια του διαχωρισμού της διαχείρισης μεταξύ των συνδρομικών υποδομών και του, των σειρμών. Αυτό θα πρέπει να το επενθυμίσουμε ότι αυτό δεν είναι λογικό και το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτρέψει το άνοιγμα στον ανταγωνισμό στο σιδηρόδρομο και ε, βοηθά να δημιουργούνται ατυχήματα αυτός ο διαχωρισμός. Εν ονόματι της μεγαλύτερης δυνατής κερδοφορίας τα Ευρω... θυσιάζουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Μπορεί να προσπαθήσετε να κερδίσετε χρόνο με την εφαρμογή σαν μόνο προπτική η αλύση των προβλημάτων τη χρήση των καλύτερων τεχνικών που υπάρχουν σε αυτή, την, αυτή τη στιγμή. Άλλη πολιτική όμω όσον αφορά του σιδηρόδρομου χρειαζόμαστε πραγματικά. Αν κάθε χρόνο έχουμε λιγότερου σιδηρομικού, λιγότερη συντηρήση, λιγότερη κατάρτιση, λιγότερε επενδύσει, αναπόφευκτα εκ νέου θα μιλάμε για ατυχήματα και θα πρέπει να εκφράζουμε συλληπιτήρια. Η πραγματική σιδηρομική ασφάλεια επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γυρίσει τη σελίδα στον ανταγωνισμό και να ανοίξει τη σελίδα τη συνεργασία. Λοιπόν, κανεί στο τέλο των συζητήσεων δεν μπορεί να αρνηθεί ποιε είναι οι ευθύνε. Όσον με αφορά, εγώ αρνούμαι να είμαι συνένοχο στη μία αλλαγή προσανατολισμού. Πέρασε ο χρόνο σα, κύριε Νά. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Φιλιπ Κλέη εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια διαπίστωση. Οι φόροι στο Βέλγιο είναι από τους πιο ψηλούς στον κόσμο. Όμως, κυρίως οι φλαμαδοί φορολογούμενοι δεν έχουν αυτά που πρέπει σαν αποζημίωση για τους φόρους που πληρώνουν. Είναι πολύ γνωστό ότι, ότι οι σιδηρόδρομοι έχουν τεράστιες καθυστερήσεις, ότι τα βαγόνια είναι φορτωμένα στις ώρες αιχμής, ότι ο εξοπλισμός είναι απαρχιωμένος, αλλά είναι χαρακτηριστικό για, την, για τους Βέλγους πολιτικούς όταν κάτι πάει στραβά, κανείς ποτέ δεν φταίει. Και άλλη φορά είχαμε ατύχημα, ένα αντίστοιχο με αυτό του Μπάζιγεμ πρόσφατα. Και πριν από εννέα χρόνια είχαν γίνει διάφορα για να βελτιωθεί η ασφάλεια. Και τελικά το σύστημα το αυτόματο, ναι, εισήχθη, αλλά όχι επαρκώς και πολύ αργά. Το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην ασφάλεια και ότι τα διάφορα συστήματα πρέπει να είναι πιο συμβατά μεταξύ τους. Αν θέλουμε πραγματικά διαλειτουργικότητα, πρέπει να περάσουμε στο ευρωπαϊκό αυτόματο σύστημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα ταλής ανάμεσα στο Παρίσι και το Άμστερνταμ περνάει από αυτά διαφορετικά συστήματα ασφάλειας. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Με την παρέμβαση αυτή του κυρίου Κλέση έκλεισε ο κατάλογος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες. Τώρα ξεκινάμε με τους συναδέρφους που μιλούν εξ ονόματός τους. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κούν έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξότιμοι συνάδελφοι. Η σύγκρουση των δύο τρένων εδώ στις Βρυξέλλες που οδήγησε σε αυτό το φοβερό δυστύχημα μας ε, έπληξε πολύ και η σκέψη μας είναι στις οικογένειες, ...τους φίλους, ε, τους συγγενείς των θυμάτων. Μετά από τέτοια δυστυχήματα Κανένα τίνει να αναζητεί τους φταίχτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, η Διατάξη Ασφαλείας. που προωθήσαμε με την οδηγία 2004-49 δεν μπορούν όμως να θεωρηθούν υπεύθυνοι. Από την άλλη μεριά έχουμε και το θέμα κατά πόσον οι διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να ενδυναμωθούν περισσότερο. Οι έρευνες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και γι' αυτό δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιο θα είναι το αίτιο του δυστυχήματος. Ε, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κάτι που ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ούτε και τεχνικό πρόβλημα. Αυτά παίζουν πάντα ένα ρόλο όταν εξτάζουμε θέματα σε των δρόμων. Και γι' αυτό όλοι οι... εκείνοι που ε, διαχειρίζονται τους σιδηροδρόμου είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν κάθε φορά κατά πόσον οι ισχύουσε διατάξει ασφαλείας τηρούνται. Εγώ δεν θέλω να σας πω τίποτα από γερμανικής πλευράς, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς στη Γερμανία προσπαθήσαμε τουλάχιστον να εφαρμόσουμε την οδηγία στο σύνολό της. Και εάν υπάρχει πρόβλημα ανθρώπινου παράδειγμα, θα πρέπει να προβλέψουμε ένα ε, τεχνολογικό ε, μια τεχνολογική λύση αν παραδείγματος κανένας περάσει από το κόκκινο φανάρι θα πρέπει αυτό με το τρένο να φρενάρει θα πρέπει όλες αυτές οι διατάξεις να εφαρμοστούν ούτως ώστε να μπορέσουμε τον έξω να παρεμβαίνουμε στην Επιτροπή Μεταφορών από κοινού θα κάνουμε την αξιολόγηση που χρειάζεται και να καταλήξουμε συμπεράσματα όσον αφορά και τι διατάξει ασφαλείας. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ο κύριο Ταραμπέλα τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η... Το ατύχημα στο Μπάζιγκαμ έξω από τι Βρυξέλλε είχε 18 θύματα και των 60 τραυματίε. Η σκέψη μα είναι στι οικογένειέ του. Δεν ξέρουμε τι αιτίε, γίνεται έρευνα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη αναχώρα μέλο, Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να ασχοληθεί με τα συστήματα ασφάλειας, σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους και αν είναι αποτελεσματικά. Η αξιολόγηση αυτή όμως της ασφάλειας στην Ευρώπη πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να συμπεριλάβει και τι συνθήκε εργασία ε, των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να υπάρξει μια αξιολόγηση τη ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων με μια γενική προσέγγιση, διότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει έρθει η στιγμή να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ελευθέρωσης και κατάργησης των κοινοφιλών υπηρεσιών, ποιος έχει αποφεληθεί, ποιος έχει ζημιωθεί. Πρέπει να συγκρίνουμε επίση τι ευρωπαϊκέ διατάξει ασφάλεια, σήμανση, τι ηθίκε εργασίε, την ελευθέρωση των σιδηροδρόμων σε κάθε χώρα μέλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να δει γενικότερα τον ρόλο των κοινοφιλών υπηρεσιών. Οι σοσιαλιστέ εδώ και καιρό ζητούν μια θετική δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε παρατέρω τι κοινοφιλεί υπηρεσίε. Είναι στοιχείο κλειδί διότι έτσι οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορέσουν να έχουν και σωστή χρηματοδότηση για να ισχύσει η οικουμενικότητα και η ισότιμη πρόσβαση όλων σε αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Yes, that's, that's right. Will Παρακαλώ. Κύριε Ταραμπέλα, δέχεστε την ερώτηση, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, μια ερώτηση στον κύριο Ταραμπέλα τον οποίον εκτιμάω ιδιαίτερα. Αλλά από την άλλη μεριά, οι βελγικοί σιδηρόδρομοι είναι αυτοί που παίρνουν τις περισσότερες επιδοτήσει στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι φταίει η ελευθέρωση. Ούτε μπορώ να δεχτώ άλλες δικαιολογίες. Μα οι σοσιαλιστές είναι εκείνοι που έχουν ιδιαίτερε σχέσεις με τα συνδικάτα των σιδηροδρόμων. Και το σύστημα αυτό των σιδηροδρόμων θα τύχει καλύτερη διαχείρισης. Κύριε Ήθελα να πω στον κύριο Έπινγκ ότι εδώ δεν συζητάμε ε, εκλογικά. Είχαμε μια καταστροφή με τα τρένα και άλλε συζητάμε για τι αιτίε. Υπάρχει μέσα στου που ποτέ δεν το ξεχνάμε, είναι ο ανθρώπινο παράγοντα. Και σε κάθε φιλελευθερωποίηση που την οποία προασπίζεται, εγώ την υπερασπίζω πολύ λιγότερο, κυρίω στι δημόσιε υπηρεσίε, βέβαια όχι, παραμελείται ένα παράγοντα. Ασκείται μεγάλη πίεση στο προσωπικό που δουλεύει ατελείωτες ώρες, όλο και περισσότερες ώρες, χωρίς ε, ανάπαυση. Και όταν είσαι μηχανοδηγός, τίθεται θέμα ασφαλείας των επιβατών και τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας και η εξέλιξή τους. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντική παράμετρο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, το φρικτό ε, συνδρομικό δυστύχημα ήταν, είναι μια τραγωδία για τι οικογένειε των θυμάτων και του φίλου του. Θα πρέπει να βγάλουμε όμω τα διδάγματα από την τραγωδία αυτή, αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να αποφύγουμε παρόμοιε ε, απώλειες στο μέλλον. Γι' αυτό η φωνή των σιδηροδρομικών πρέπει να ακουστεί και να εισακουστεί. Δεν είναι ασφαλή τα τρένα και για του εργαζόμενου και για του επιβάτε. Είναι απαράδεκτο να ακούμε έναν Βρετανό τόρι ευρωβουλευτή να στυλιτεύει τους Βέλγους για αυτό που είπαμε. Ενώ αυτό προέρχεται από άρση της νομοθεσίας και φιλελευθεροποίηση. Αυτό κατέφερε μεγάλο πλήγμα στους ιδεοδρόμους ως δημόσια υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι σιδηροδρομικοί στο Βέλγιο είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Το βλέπουμε αυτό από αυθόρμητες απεργίες στους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους μέρες αμέσως μετά την τραγωδία και είναι το τρίτο σοβαρό δυστύχημα μέσα σε εννέα μήνες στο Βέλγιο. Στην προηγούμενη τραγωδία το 2001 στο Βέλγιο υποσχέθηκαν ότι θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας, δεν έγιναν. Και οι σιδηροδρομικοί στο Βέλγιο είναι που συνεχίζει να δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες με όλο και λιγότερα διαλύματα. για ανάπαυση αυτό σημαίνει λιγότερη ασφάλεια και φυσικά η ύπουλη πολιτική της Κομισιόν για φιλελευθερωποίηση και άρση της νομοθεσίας ε, είναι απειλή για την ασφαλειά τους. Είναι πίεση στις επιχειρήσεις. Η καλύτερη εγγύηση είναι η συνδρομική υποδομή να παραμείνει υπό το δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο και με αναγκαίες επενδύσεις. Ευχαριστώ. κύριος Μπαχ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στι οικογένειε. Βέβαια, δεν θα του ε, παρηγορήσει πάρα πολύ όταν τονίζουμε ότι οι συνδρόμοι εξακολουθούν να είναι από τους πιο σίγουρα, πιο σίγουρα μεταφορικά μέτρα και ότι ο αριθμό των δυστυχημάτων είναι χαμηλό. Γιατί βέβαια οπωσδήποτε τίθεται το θέμα πώ μπορέσαμε να ζήσουμε αυτή την καταστροφή. Ή τεχνικοί εμπειρογνώμονες και μετά τα δικαστήρια θα εξετάσουν το θέμα. Εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο ήταν το σφάλμα μέχρι στιγμή στην ε, προετοιμασία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια δυστυχήματα στο μέλλον. Γιατί κάθε δυστύχημα είναι ένα περιττό δυστύχημα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να τονίσω κάποια θέματα που έχουν επιτρέψει στην ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις των σιδερόμων, αντί να τους θέσουμε εκ μιας αρχής σε ανταγωνισμό, έπρεπε να υπάρχει πρώτα μια τεχνολογική εναρμόνιση. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει στη δεκαετία του 90 που τα τόνισε και ο κύριος Κάλλας. Και μόνο μετά από εναρμόνιση θα μπορούσαμε να είχαμε ε, ανταγωνισμό. Γιατί ο κατακρισμός της αγοράς σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα ε, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Και γι' αυτό έχω να σας πω ότι έχουμε μια κοινή ευθύνη. Αφενός δηλαδή τα κράτη-μέλη, οι επιχειρήσεις των συνδρόμων και εκείνοι που έχουν στη διαχείρισή τους την, ε, την υποδομή και η Κομισιόν επίσης θα πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση όμως έγινε μόλις πρόσφατα. Οι επιχειρήσεις των Συνδρομών δυστυχώς επέλεξαν εσφαλμένη στρατηγική. Περίμεναν πολύ καιρό ευρωπαϊκό ε, σύστημα. Ε, έκαναν πάρα πολλές εξοικονομήσεις. Επιδεινώθηκε έτσι ε, το επίπεδο του προσωπικού. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα. Θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για να μπορέσει να προωθηθεί ο εξοικονομισμό που έχει προβλεφθεί. Η κυρία Τικάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ είναι συνήθω πιο ασφαλεί, πιο γρήγορε και ρηπαίνουν λιγότερο από ό,τι οδικέ. Παρ' όλα αυτά όμω, το 2007, περίπου 2.600 άτομα υπήρξαν ε, θύματα συνδρομικών ατυχημάτων και φέρος είχαμε περισσότερα ε, τέτοια δυστυχήματα και με ε, τρένα που μεταφέρουν φορτία. Το τα ατυχήματα στο Βέλγιο με 200 τόσου νεκρού μα θυμίζουν πώ επίκαιρο το θέμα αυτό. Δυστυχώ, η οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση επιδίνωσε τι οικονομικέ δυσκολίε των διαχειριστών των συνδρομικών επιχειρήσεων. Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού υπάρχει έλλειψη πόρων προκειμένου να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα. Και αυτό είναι μία από τις αιτίες του δυστυχήματος και χιλιάδες διαδρομικοί χάνουν τις δουλειές τους. Καλό ότι τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να πάρουν μέτρα. Πρώτον, να αποκατασταθεί η υποδομή στους σιδηροδρόμους και στο σιδηροδρομικό υλικό, έτσι ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική μεταφορά με τους σιδηροδρόμους και δεύτερον να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και τρίτο, νέα υποδομή και συστήματα RTMS. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάντσιαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα πρόσφατα συνδρομικά δυστυχήματα που έπληξαν την Ευρώπη, χθε στην Ιταλία, σήμερα το Βέλγιο, μα επιβάλλουν να σκεφτούμε πού πάσχει το σύστημα και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθούν οι παροχέ όσον αφορά την ασφάλεια. Παραδείγματο χάρη είναι περίεργο το ότι η Ένωση ήδη το 2001 επεξεργάστηκε ένα σύστημα για την υποπτία τη ιδρομικών μεταφορών, τα δίκτυα RDMS, και όμω έχουν περάσει 10 χρόνια και το σύστημα από ελάχιστε χώρε έχει υιοθετηθεί. Ακόμα υπάρχουν στην Ένωση πάνω από 20 διαφορετικά συστήματα σιδηροδρομική ασφάλεια. Είναι προφανέ ότι αυτό δημιουργεί δυσκολίε ιδιαίτερα στις διεθνείς διαδρομές. Η προσαρμογή λοιπόν της υποδομής και του ισοδοδομικού υλικού απαιτεί αξιολόγηση και προσαρμογή οικονομικής και τεχνικής μορφής και πρέπει φυσικά αυτά να τα διαχειριστούν οι επιχειρήσεις. Επισημένω όμως ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν ορίζει προθεσμία για την προσαρμογή των εθνικών συστημάτων στα δίκτυα RTMS ζητάει από τα κράτη, μάλλον δίνει στα κράτη-μέλη την αρμοδιότητα αυτή να αξιολογήσουν τα, το σιδηροδρομικό υλικό. Καλό θα είναι να οριστεί η ημερομηνία ή να δοθούν κίνητρα για τι επενδύσει ή να αφαιρεθούν κίνητρα από αυτού, να αφαιρεθούν επενδύσει, μάλλον από αυτού που δεν προσαρμόζονται από αυτού που δεν χρησιμοποιούν τα συστήματα. Κάτι άλλο. Δεν πρέπει να επιβραδυνθεί η διασύνδεση και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς έχουμε ένα εθνικό όργανο ανεξάρτητο για την ασφάλεια που θα ελέγξει ε, κατά πόσο είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν τα συστήματα ασφαλείας. Πρέπει να επιμείνουμε να δίνονται πιστοποιητικά ασφαλείας ως προϋπόθεση προκειμένου να δίνεται άδεια άσκησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή απελευθερωμένη στη αγορά με ενισχυμένο σε κεντρικό επίπεδο οι εξουσίες του αρμόδιου οργανισμού για τους ελέγχους. Ευχαριστώ. Η κυρία Σερατσάνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Μετά το πρόσφατο δυστύχημα στις Βρυξέλλε, που πολλοί συνάδελφοι μα το θύμισαν για μια φορά οι προβολείς στράφηκαν στην ασφάλεια στα τρένα. Η οδηγία 2004 για την ασφάλεια για τα τρένα γενικά ορίζει ότι οι επιχειρήσει και οι αρμόδιοι φορεί για την υποδομή είναι συνυπεύθυνοι για την ασφάλεια. Ο καθένα στι αρμοδιότητέ του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του συγκεκριμένου δυστυχήματο στο Βέλγιο φαίνεται ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθο. Βέβαια θα περιμένουμε τι ανακρίσει, αλλά το τρένο φαίνεται ότι δεν είχε αυτόματο σύστημα τροχοπέδηση. Η Κομισιόν γνωρίζοντα ε, τι συμβαίνει, ότι δηλαδή το όργανο αυτό ασφάλεια δεν το έχουν πολλέ χώρε. Η Κομισιόν, λέω, σκοπεύει να κινήσει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε σε όλο το Δίκτυο της να υπάρχει αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίτρας για δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων αυτού του ατυχήματος. Κατά δεύτερο λόγο, να σας αναφέρω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα συζητούμε και είναι θετικό το ότι συζητούμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μια αγορά που έχει υποστεί την απελευθέρωση λειτουργεί καλύτερα από το να υπάρχει μόνο κάποια κριτική εταιρεία. Όμως τώρα το θέμα δεν είναι μόνο η κυριότητα του δικτύου για της εταιρεία. Το θέμα είναι η αγορά. Η αγορά είναι ελεύθερη, είναι μια ρυθμισμένη και κατευθυνόμενη αγορά. Αλλιώς πάμε σε μοντέλο μονοπωλιακό. Πολύ συχνά έχουμε ως εξή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικά συστήματα και πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν περισσότερα από ένα συστήματα ασφαλείας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα τεχνητό φραγμό στην εταιρεία που διεκδικεί μονοπωλιακή θέση στην αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις δε, δεν ε, υιοθετείται κάποια αλλαγή, καινούριο υλικό, ε, ακριβώς για να παρεμποδιστεί η ανέλυξη του ανταγωνιστή. Να γιατί προκύπτουν προβλήματα ασφάλειας. Και αν δείτε ως γίνεται η κατανομή των ε, διορθωτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη θα διαπιστώσετε ότι ουσιαστικά για υποδομές υδροδρομικές δεν δίνονται χρήματα. Αιτήσει οι οποίε προσκρούν στο κενό, στην διαφορία. Το συμφέρον επομένω είναι αυτών που είναι και καθιδρυμένοι, ε, έχουν ήδη κάποια θέση στην αγορά, να μην θέλουν να έρθουν καινούργια, να, να μην υπάρχει ανταγωνισμό, μην έρθει κανεί από άλλο κράτο μέλο. Και βλέπουμε επομένω ότι τελικά ε, ε, χαμένο βγαίνει ασφάλεια. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, τα γεγονότα του Μπάζιγκεν συνεκλώνησαν και εμάς και όλους τους Ευρωπαίους και θα πρέπει επομένω να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα και θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια πιο μακρόπνοη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Είπαμε ότι ακόμα στο Βέλγιο δεν έχουμε το αυτόματο σύστημα πέδησης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μείνει τα χέρια σταυρωμένα. Το αντίθετο, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε κάποια δική τη μελέτη αξιολόγηση και να δώσει κάποιε απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Φερρυπίν, οι εταιρείε ακόμα και ιδιωτικέ απαιτείται από το 2013 να βάζουν σε, όλα τους τα, όλους τους, τους συρμούς το σύστημα αιτίας. Και, Πρόεδρε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το σύστημα ασφάλειας βρίσκεται μόνο εγκατεστημένο σε 800 χιλιόμετρα στο δρομικές γραμμές, ενώ στο Βέλγιο μόνο έχουμε 3.000 και χιλιόμετρα γραμμές. Άρα βλέπουμε ότι ο εξοπλισμός είναι ανεπαρκής και άρα χρειαζόμαστε περισσότερη πλαισίωση. Άρα να κάτσουμε και να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει περισσότερη πίεση, γιατί υπάρχει πίεση λόγω του ανταγωνισμού. Άρα να κάτσουμε και να δούμε πώς θα καθορίσουμε και περισσότερα περιθώρια ε, ανάπαυσης, χρόνου ανάπαυσης, χρόνου εναλλαγή για του οδηγού, όπω κάναμε και για τα φορτηγά, θα πρέπει να να κάνετε μια αξιολόγηση και να καταλήξετε κατά, κατά πόσο έχουμε την πολιτική να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Ο κύριο Κρέιμερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το φοβερό δυστύχημα έλαβε χώρα όταν δύο ε, με, μεταξύ δύο σιδηροδρόμων στο εθνικό δίκαιο, στο κρατικό δίκαιο, ε, ε κρατικές ε, δεν υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός. Ο κύριος Γκρός είπε ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει η τεχνολογία σύμφωνα με την οποία εάν κανένας δεν σταματήσει στο κόκκινο αυτόματα τροχοπεδείται το τρένο. Γιατί δεν είχε ε, εγκατασταθεί αυτό το, αυτό το σύστημα. Μη συζητήσει για το RTMS. Αυτό είναι για το μέλλον. Αυτό δεν απαλλάσσει όμως κανένα να εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο. Είναι εθνικό έργο. Γιατί το Βέλγιο εδώ και 20 χρόνια δεν επένδυσε στην ασφάλεια. Α μην είχαν φτιάξει κανένα δύο χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο παραπάνω. Α είχαν χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα ασφαλεία και να μην υπάρχουν αυτά τα δυστυχήματα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαμε ένα τέτοιο δυστύχημα. Δεν έχω άλλο ομιλητή για το ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Υπάρχει κάποιος άλλος που επιθυμεί να μιλήσει. Όχι. Επομένως, περνάμε εξ ονόματος της Επιτροπής στον Επίτροπο τον κύριο Κάλλας. Thank um, Κάλλας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και η σημερινή συζήτηση έχει αφορμή το τραγικό αυτό ατύχημα που έλαβε χώρα στο Βέλγιο. Κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστα δεμένο με τις εξελίξεις στην ασφάλεια των μεταφορών στην Ευρώπη. Και έτσι εμείς εκπονούμε αυτή τη λευκή βίβλο και λαμβάνουμε σοβαρά όλες αυτές τις πτυχές του θέματος. Και φυσικά, όπως αναφέρθηκε τόσες φορές, ο σιδηρόδρομος είναι ένας ε, ασφαλής τρόπος μεταφοράς παρόλα αυτά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τη συνέχεια θα έχει το λεγόμενο πρώτο, παγιό, για την πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Το δε σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη έχει σχεδιαστεί, ούτως ώστε να είναι διαλειτουργικό και βεβαίω είναι αξιόλογο σύστημα ε, περιέχει κάποια σοβαρά στοιχεία ασφάλειας αλλά ακόμα η ασφάλεια είναι αρμοδιότητα εθνική πέραν των συστημάτων αυτό το ε, σύστημα για το DMS είναι μια ιδέα που την έχει οθετήσει το σύστημα διαχείρισης εν του ορίζοντα του 2020 και θέλουμε ε, να καλύψουμε μέχρι τότε περί τα 2.000 χιλιόμετρα γραμμής και να καλύψουμε και το Βέλγιο. Γίνονται σημαντικές επενδύσεις. Επομένως έχουμε πολλούς πόρους οι οποίοι κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση και για το σύστημα αυτοπαίδησης, το αυτόματο. Αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ θετικό το ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί και θα μας στηρίξει. Πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως, πάντοτε είναι σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας και το πιο σημαντικό πέραν των προτύπων είναι το να να αλλάξουμε κάποια, κάποιες ε, υποδομές που είναι εκεί από το 19ο αιώνα. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε για τον ανθρώπινο παραγόντα ότι ποτέ 100% δεν είναι ε, αδύνατο να υπάρξει ανθρώπινο σφάλμα. Τώρα άλλη μια παρατήρηση για την απελευθέρωση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Κανείς δεν μπορεί να ε, εμποδίσει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν κάποιες ε, δημόσιες υπηρεσίες όσο και αν υπάρχει απελευθέρωση. Επομένως, η απελευθέρωση δεν σημαίνει αποκλεισμό των, ε, της καλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Έληξε. Οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν σε πέντε λεπτά ακριβώς.